για την ψηφοφορία για το ICI για την έκθεση του κυρίου Ντέβα. Άκουσα ότι στην Επιτροπή Ίντα υπάρχει, γίνεται μια συζήτηση σχετικά με το εάν όντως υπάρχει ε, νόημα να γίνει ψηφοφορία επί της εκθέσης αυτής, διότι πρόκειται να την παραπέμψουν εκ νέου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θεωρώντα ότι η νομική βάση τώρα με τη συνθήκη τη Λισαβόνα δεν είναι πια η σωστή. Μάλιστα, λέει η Πρόεδρο, θα το, θα το πω αυτό σε λίγο. Πάντω, τώρα, για τη γνωμοδότηση του κυρίου Ντέβα για την αναθεώρηση του μηχανισμού συνεργασία με τις εκβιομηχανισμένες χώρες. Επειδή ε, θα τεθεί σε ισχύ η συνθήκη της ε, Λισαβόνας από 1η Δεκεμβρίου, η αρμόδια επιτουσίας επιτροπή δεν προτίθεται να ψηφίσει επιτουσίας. Διότι η νομική βάση που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν υφίσταται πλέον ε, υπό τη νέα συνθήκη. Θα χρειαστεί λοιπόν να γίνει νέα πρόταση για τον μηχανισμό ICI. Άρα η διαδικασία θα πρέπει να αρχίσει εκ νέου, πιθανώς σε διαδικασία συναπόφασης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ακόμη ωστόσο δεν έχουμε ε, σαφείς πληροφορίες από την αρμόδια επιστουσίας επιτροπή για το πώς επιθυμεί να προχωρήσει. Ο εισηγητή λοιπόν της ε, Επιτροπής Ανάπτυξης προτείνει να ε, συνεχίσουμε να κάνουμε την ψηφοφορία ώστε να επιβεβαιώσουμε την θέση μα για το θέμα και ιδίω για την χρηματοδότηση τη ICI. Οι θέσει που θα λάβουμε σήμερα βεβαίως δεν μας δεσμεύει εάν και εφόσον προ, ε, ε, μας ζητηθεί να επανεξάσουμε το θέμα. Συμφωνείτε με τη διαδικασία αυτή καλά. Συμφωνείτε λοιπόν, έχει καλώ προχωρούμε τότε στην ψηφοφορία. Η τροπολογία υπαριθμών 2 πρώτα. Παρακαλώ υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται και αυτή. 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 5 υπέρ. κατά αποχές εγκρίνεται ζητείτε ψηφοφορία κατά τμήματα για την τροπολογία 6 πρώτο τμήμα παρακαλώ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 1 του εισηγητού. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η γνωμοδότηση στο σύνολό της όπως τροποποιήθηκε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα οι τροπολογίες για τον μηχανισμό σταθερότητας. Τροπολογία 1. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Η γνωμοδότηση στο σύνολό της παρακαλώ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται και αυτή. Άρα έληξε το θέμα υπαριθμών 15. Χάσαμε μισή ώρα περίπου σε συζητήσεις με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Συμφωνία Κοτονού, για την αναθεώρηση της Συμφωνίας Κοτονού Γι' αυτό προτείνω να μην παρουσιάσω την έκθεσή μου ε, σε εσά, αλλά να σας προσκαλέσω ευθύ αμέσω να θέσετε ερωτήσεις, εάν έχετε κάποιες. Συμφωνείτε? Ωραία λοιπόν. Ε, δίνω την ε, δυνατότητα να λάβετε το λόγο για να θέσετε ερωτήσεις. Υπάρχει μια προθεσμία για κατάθεση τροπολογιών που προβλέπεται για τις 19 Νοεμβρίου την 6η απογευματινή. Αν λοιπόν δεν έχετε ερωτήσεις μπορείτε ωστόσο πάντοτε να γράψετε τις ε, τροπολογίες σας και να τις υποβάλλετε. Κύριε Χάλεμ Ντεζίρ. Πρόεδρε, εννοείται ερωτήσεις προς εσάς την ίδια ως εισηγήτρια ή σχόλια, παρεμβάσεις. Ωραία. Καταρχάς, να πω ότι έλαβα γνώση της έκθεσης, του σχεδίου έκθεσης με ιδιαίτερο ενδιαφέρον νομίζω ότι πραγματικά αντικατοπτρίζει τις βασικές ανησυχίες που εκφράστηκαν και στην Επιτροπή μας στις πρώτες ανταλλαγές απόψεων που είχαμε. Να σας πω λοιπόν ότι η ομάδα μου θα προσφέρει την ε, στήριξή της στην ε, παρουσίαση που κάνετε των προκλήσεων. Όπως το ανέφερα και κατά την ανταλλαγή που είχαμε προηγουμένως με την Επιτροπή και που σε ένα σημείο που εσείς καλύπτετε στο τέταρτο σημείο της έκθεσής σας. Νομίζω οι εμπορικέ σχέσεις, ο εμπορικό τομέα θα παραμένει μια σημαντική μέρημνα. Ακόμη και αν οι συμφωνίες εταιρική σχέσης υποκαθιστούν το προηγούμενο εμπορικό καθεστώς, στις διατάξεις του άρθρου 37 των συμφωνιών Κοτονού, τώρα υπήρχε μία επιλογή που ελεύθερα μπορούσαν να διαλέξουν οι χώρε ΑΚΕ. Είτε δηλαδή να προσχωρήσουν στη Συμφωνία Κοτονού, είτε να διαλέξουν ένα άλλο εμπορικό καθεστώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μα λέει ότι τώρα δεν θα υπάρχει πλέον επιλογή. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι η προσχώρηση στι συμφωνίε εμπορική σχέση είναι υποχρεωτική. Διαφορά σε σχέση με, τι ε, με την μορφή που είχαν ω τώρα οι συμφωνίε Κοτονού. Όταν βλέπουμε τι δυσκολίε υπάρχουν να συμπέσουν τα πλαίσια των ε, συμφωνών οικονομικής σχέσης με τις ιδιαίτερες ανάγκες που υπάρχουν, ειδικά στην Αφρική, εδώ υπάρχει μάλλον ένα μικρό πρόβλημα. Δεν μπορούμε να, να αποκλείσουμε την περίπτωση κάποιες χώρες να περνάνε σε συμφωνίες οικονομικής σχέσης, ακόμη και αν υπάρχουν διάφορες μορφές εμπορικής ε, συνεργασίας με την Ευρώπη. Δεν μπορούμε να αρνηθούμε να μην υπάρχει καμία ιδιαιτερότητα στι εμπορικέ σχέσει μεταξύ των χωρών ΑΚΕ και τη Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια των συμφωνιών Κοτονού. Εδώ νομίζω ότι υπάρχει ένα θέμα και έχει δίκιο η κυρία Ζολή που το τονίζει στο σχέδιο εκθεσή τη. Θα πρέπει αυτό να διορθωθεί. Και ίσω σχετικά θα πρέπει να υποβληθούν και τροπολογίε. Για τι άλλε μεγάλε προτεραιότητε, κλιματικέ ε, αλλαγέ, κάτι που ήδη συζητάτε, ή την ε, τη στήριξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργεια, έπειτα την επισητιστική κρίση, την επισητιστική ασφάλεια, την ε, αγορά αεροτρέων γεών, τον εξοπλισμό, τον γεωργικό εξοπλισμό που χρειάζεται. Ε, όλα αυτά τα παρουσιάζεται πολύ σωστά, αλλά νομίζω ότι στι διαπραγματεύσει αυτέ για την αναθεώρηση των συμφωνιών Κοτονού θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση σε όλα αυτά. Βεβαίω η ανάπτυξη, η αναπτυξική βοήθεια, η διαφοροποίηση του τομέα τη οικονομία, η εισαγωγή των υπηρεσιών, ο οικοβιομηχανισμό όπου είναι δυνατόν, οι υποδομέ είναι σημαντικέ. Αλλά δεν υπάρχει ανάπτυξη και μα το έδειξε αυτό η επιστημιστική κρίση χωρί γεωργία. Αν οι γεωργοί δεν αμείβονται σωστά, αν δεν έχουν τι δυνατότητε να καλύπτουν τι ανάγκε, τι διατροφικέ του πληθυσμού. Θα ήθελα λοιπόν στη συζήτηση που θα έχουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο να προβάλλουμε και αυτό το επιχείρημα. Για τα προβλήματα των ανθρώπινων δικαιωμάτων τα έχουμε αναφέρει, αλλά εδώ θα πρέπει να κάνουμε ένα συσχετισμό με τη διαφάνεια, με την καταπολέμηση τη διαφθορά, με την καταπολέμηση τη φοροδιαφυγή. Και πάλι τα πρόσφατα γεγονότα, ε, αναφερθήκαμε προηγουμένω στην Γουινέα, μια χώρα με εξαιρετικού πόρου μεν, αλλά δεν θα επιτελέσει πρόοδο, ούτε θα επιτελέσουμε γενικώ πρόοδο στην ε, ε, στα ανθρώπινα δικαιώματα, ούτε στην ανάπτυξη και την οικονομία, αν δεν ε, εκδημοκρατιστούν οι χώρε αυτέ. Να λοιπόν, ε, πώ θα πρέπει να διαρθωθούν όλα αυτά τα θέματα και να το συνδυάσουμε αυτό και με κάτι που σα είναι προσφυλέ, κυρία Πρόεδρε, με τη φοροδιαφυγή και την όλη προσπάθεια να καταπολεμήσουμε την χρηματοπιστωτική κρίση. Να λοιπόν, κάποια σημεία που θα έπρεπε να τονιστούν, αλλά σε κάθε περίπτωση το περιεχόμενο τη πρότασή σα μα βρίσκει απόλυτα σύμφωνο. Σα ευχαριστώ, κύριε Κάσμαν. Thank you. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ. Και ανέφερε κάτι το οποίο με απασχόλησε και εμένα, δηλαδή το θέμα των ε, δικαιωμάτων των μειονοτήτων στα πλαίσια της ε, Συμφωνίας Κοτονού, διότι πολύ συχνά οι σχετικές ρήτρε έχουν αγνοηθεί και τα σχετικά με τους ομοφιλοφίλους οι οποίοι υφίστανται επιθέσεις. Είδαμε και στο Μπουρούντι πως ε, είχαμε την ποινικοποίηση της έκφρασης των σεξουαλικών προτιμήσεων στη δενιγυρία έχει επιβληθεί η θανατική ποινή. Οπότε δεν μπορώ να συμφωνήσω με τα όσα είπε ο κ. Ντεζίρ. Merci, Monsieur s'il vous plaît. Euh, Και εγώ, κυρία Πρόεδρε, να σας πω για την έκθεση ότι θεωρώ ότι πρόκειται για ένα κείμενο ενδελεχές το οποίο αντιστοιχεί ε, στην ε, πρόκληση της αναθεώρησης της Συμφωνίας Κοτονού. Πρόκειται για ένα πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο όμως υπάρχουν διάφορες ε, ε αλλαγές, οπότε πρέπει να κατεβάσουμε κάποιες τροπολογίες και πρώτα πρώτα όσον αφορά το Δέλτα, την τελική παράγραφο Δέλτα εκεί που λέει ότι προβλέπει την περιφερειοποίηση της ΑΣΕΠ εδώ είναι προβληματικό αυτό γιατί εκεί που λέει η επιτελικό αναπόφευκτο αυτό οδηγεί στο ότι η περιφερειοποίηση είναι κάτι το κακό Πρέπει επίσης να δούμε τη διαφοροποίηση που προβλέπετε εδώ και που τα διάφορα όργανα για τις υπηρεσίες που εμπλέκονται, οπότε θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τα καινούργια όργανα της ε, ΑΚΕΙ στα πλαίσια της Συμφωνίας Κοτονού. Οπότε θα πρέπει να δούμε πώς θα παραμείνει όσα έχει η Δέλτα. Η παράγραφος Δέλτα. Και λέει εδώ πέρα για τους φορείς κοινωνίας των πολιτών, στα πλαίσια σκοτωνού επομένω. Να δούμε πώ είναι δυνατόν η κοινωνία των πολιτών να μπορεί να δραματίσει ένα σημαντικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί δεν είναι δυνατόν να θεωρήσουμε ότι αυτοί οι φορεί είναι το ίδιο σημαντικό όσο τα εθνικά κοινοβούλια. Οι φορεί τη κοινωνία των πολιτών επίση θα πρέπει να δούμε πώ θα χαρακτηριστούν σε σχέση με την ιδεολογική έκθεση. Γιατί το κοινοβούλια, το εθνικό, το, το, η σωμερή συνέλευση δεν εκλήθησαν να διαβουλευτούν όσον αφορά την, ε, την διαπραγματευτική εντολή. Τώρα, στο ΓΑΜΕ, τελευταία φράση έχει πολύ ότι απευθύνει μια έκκληση να υπάρχει ένας υποχρεωτικός μηχανισμός που να υποχρεώνει τις πολυεθνικές να φορολογούνται ε, επί των κερδών τους σε κάθε χώρα και θα πρέπει επομένω αυτό να εφαρμοστεί από τον ΟΗΕ για όλες τις πολυεθνικές. Τώρα, στην παράγραφο 13. Το δεύτερο τμήμα είναι προβληματικό ιδίω η αγγλική εκδοχή. Το δικαίωμα του πληθυσμού να ελέγχει τις γεωργικές γης κάτι το οποίο δεν συμβαδίζει με την οικονομία της αγοράς στην παράγραφο 15 τα Εθνικά Κοινοβούλια γιατί θα πρέπει να τονίσουμε ότι χρειάζεται να δούμε τι θα γίνει σε αυτή την πολιτική διάσταση, διότι έχει ξεχαστεί η πολιτική πτυχή του θέματος. Χρειάζονται σημαντικές μεταρρυθμίσεις και είναι πάντοτε επίκαιρες και άρα θα χρειάζεται να γίνει εδώ μία παράγραφος να προσθεθεί. σε ΠΕΗ θα πρέπει να απευθυνθεί στον ασκούντα την Προεδρία του Σουδάν και να δούμε πώς θα καλυφθεί και αυτό το θέμα από τη συμφωνία. Ευχαριστούμε που πήρατε το λόγο και θα ήθελα να σας πω, Λεπρόεδρος, ότι βεβαίως όλα τα θέματα της Συμφωνίας Κοτονού δεν καλύπτονται από το σχέδιο κειμένου γιατί έχουμε περιορισμό όσον αφορά το μέγεθο τη έκθεση. Οπότε όλα αυτά θα καλυφθούν με τι τροπολογίε που θα λάβουμε υπόψη. Και τώρα το λόγο έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα είμαι πολύ σύντομο, κυρία Πρόεδρε για αυτά τα θέματα τα οποία αφορούν εμά, αλλά πρώτα πρώτα συγχαρητήρια για την έκθεση διότι είναι εξαιρετική αυτή η ανάλυση του πλαισίου και των θεμάτων τα οποία σας απασχολούν εμείς συμφωνούμε με τα περισσότερα από όσα διατυπώνεται. Και φάνηκε και από τη συζήτηση ότι τα περισσότερα θέματα καλύπτονται από την διαπραγματεύση που βρίσκεται να εξελίξει. Το μόνο θέμα το οποίο μας απασχολεί κάπως είναι αυτή η αναδιανομή της γης Εδώ είναι λίγο δύσκολη η ρυθμίση γιατί η γεωργική πολιτική στην οποία αναφέρει ο κ. Ντεζίρ πρόκειται να καλυφθεί από τις συζητήσεις και επαφές που θα γίνουν και περιμένουμε τις προτάσεις της ομάδας ΑΚΕ. Εμείς δεν έχουμε κάνει προτάσεις. Να δούμε τι θα γίνει όσον αφορά την περιφερειακή ολοκλήρωση. Εκεί θα κατέθεσαν κάποιες προτάσεις. Όσον αφορά δε την ε, διαφθορά, είναι το κείμενο και το μόνο το οποίο μπορούσαμε να ε, προσθέσουμε είναι η χρηστική κυβέρνηση όσον αφορά τα φορολογικά. Η πρότασή μας επομένως αφορά ακριβώς μια πιο σωστή φορολογική πολιτική το οποίο έχει να κάνει ακριβώς με το θέμα το, της μεσονομικής πολιτικής και της φορολογικής πολιτικής. Τώρα, αφορά αυτό το οποίο είπε ο κ. Κάσμαν κατά των δυσμενών διακρίσεων, προτείναμε για το άρθρο 8 να αντικατασταθεί η σχετική ρήτρα και να μπει η ρήτρα, η αντίστοιχη, τη συνθήκη τη Λισαβόνα που είναι πιο ολοκληρωμένη και που αναφέρεται ρητό στα θέματα που αναφέρατε Να δούμε όμω εάν και ο πλευρά ΑΚΕ αυτό θα γίνει αποδεκτό. Αυτό το πήρε ο κύριο Πρέντα. Κυρίω όσον αφορά την εμπλοκή τη κοινωνία των πολιτών. Δεν είναι εταίρος, δεν είναι συμβαλόμενος η κοινωνία των πολιτών. Προβλέπεται όμως η εμπλοκή της κοινωνίας των πολιτών. Οπότε θα πρέπει να βρεθεί το μέσο, το ώστε να δοθεί η δυνατότητα προς τούτο. Θέλουμε μέρος να γίνει ένας δομημένος διάλογος με την κοινωνία των πολιτών και να καλύψουμε όλες τις πτυχές της ε, αναπτυξιακής πολιτικής ούτως ώστε να δούμε και με τι μηχανισμούς θα μπορέσουμε να συνδέσουμε με την υπόθεσή μας στην κοινωνία των πολιτών ακριβώς όπως έγινε σήμερα το πρωί με την Επιτροπή. Οπότε έχει γίνει ενημέρωση της ΟΚΕ και της ε, Σουμερού Συνέλευσης. Επίση, Επίσης, θα πρέπει να σας τονίσω ότι αυτή είναι θεώρηση. Είναι τεχνοκρατικού, τεχνικού χαρακτήρα. Δεν αφορά την ουσία της συμφωνίας. Άρα θα πρέπει κάποια στιγμή να γίνει μια πολύ βρετερή διαβούλευση. Βέβαια, έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μέχρι να λήξει η συνθήκη του 2020. Άρα, θα συνεχίσουμε γίνοντας σε αυτό το ζωντανό πλαίσιο, που είναι αποτελεσματικό, στον πρώτη σχέση μας με τις χώρες εκείνες. Ευχαριστώ. Να κλείσουμε τη συζήτηση αφού δώσουμε το λόγο και στον κύριο Ντέβα γιατί εφόσον η συζήτηση έχει κλείσει κανονικώς έχετε το λόγο για 45 μόνο δευτερόλεπτα. Πολύ σύντομα, Πρόεδρε, έχουμε μια πολύ στενή σχέση με τις χώρες εταίρους που έχουν ε, απέναντί μας κάποιο χρέος. Γιατί δεν είμαστε τόσο αυστηροί με τις χώρες με τις χώρες που έχουν ε, προβλέψει τη θανατική ποινή. Να σας θυμίσω την ημερομηνία της 19ης Νοεμβρίου στις 6 το απόγευμα για να αποστείλετε τις τροπολογίες σας για την έκθεση αυτή. Περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο μηχανισμός χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας. Αυτή είναι και η βασική μας έκθεση για σήμερα. Ο κανονισμός προβλέπει αναθεώρηση ενδιάμεση για όλη τη, συνολική διάρκεια του μηχανισμού. Μια παρόμοια διαδικασία προβλέπεται για το μέσο σταθερότητα και το μηχανισμό και εκδημοκρατισμού και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η αναθεώρηση των ε, μηχανισμών θα πρέπει να ολοκληρωθεί πριν ξεκινήσουν οι συζητήσεις, εάν γίνεται, για το καθεστώς των συμφωνιών υπό αυτό το μηχανισμό. Γι' αυτό έχουμε προβλέψει ένα χρονοδιάγραμμα που θα μας επιτρέψει να ψηφίσουμε στην επόμενη έκτακτη συνεδρίασή μας στις 23 Νοεμβρίου στο Στρασβούργο. Να δώσω το λόγο στον εισηγητή, τον κύριο Μίτσελ, για να μας παρουσιάσει τις τροπολογίες που προτείνει για την έκθεση αυτή και να σχολιάσει τις πιθανές αλλαγές που θα προκύψουν από τη θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας. Κύριε Μίτσελ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τρεις παρατηρήσεις θέλω να κάνω εδώ και τα περισσότερα από τα σχόλιά μου περιλαμβάνονται στο επεξηγηματικό σημείωμα. Πρώτα απ' όλα θα θέλαμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σεβαστεί την νομοθεσία, η οποία αυτή τη στιγμή δηλώνει επισήμω ότι η ενδιάμεση αναθεώρηση πρέπει να σεβαστεί την ε, θέση σε ισχύ του μηχανισμού χρηματοδότηση τη αναπτυξιακή συνεργασία τα πρώτα τρία χρόνια λειτουργία του. Εδώ βρισκόμαστε στα δύο πρώτα χρόνια λειτουργία. Γι' αυτό μιλάμε για ενδιάμεση αναθεώρηση. Η υλοποίηση ω τώρα του ε, μηχανισμού πρέπει να γίνει με τρόπο ενεργό και κυρίω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να συμμετάσχουν πιο ενεργά. Είναι κάτι που το έχω επισημάνει και στο παρελθόν. Και εδώ υπάρχει και το θέμα του νομοθετικού κειμένου, του ιδρυτικού κειμένου του μηχανισμού χρηματοδότηση. Κάτι που για άλλη μια φορά εξέτασε με πολύ αυστηρότητα η δική μας ε, Επιτροπή και παρακολουθεί την υλοποίησή του από την θέση του σε ισχύ το 2007. Ασκήσαμε το δικαίωμα ελέγχου και βάσει τη διαδικασία τη Επιτροπολογία, αλλά εδώ δημιουργήθηκαν δυσκολίε και διαφωνίε σε σχέση με τον τρόπο που υλοποιήθηκε ο μηχανισμό και την ερμηνεία από την πλευρά τη Επιτροπή σε κάποιε από τι βασικέ διατάξει. Ωστόσο, δεν βρήκαμε σοβαρέ τι λειτουργίε ε, στην ε, ίδια την υλοποίηση του μηχανισμού στην κοινοβουλευτική μας θητεία θα χρειαστεί να ξεκινήσουμε και διαπραγματεύσεις για την μηχανισμό που θα διαδεχτεί το σημερινό. Ο μηχανισμός αυτός θα εκπνεύσει το 2013 και τότε θα πρέπει να έχει προβλεφθεί ο επόμενος. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε την ουσία και τις προτεραιότητες και να μην επιβαρύνουμε όλη αυτή τη διαδικασία με περιττέρω βασικές αλλαγές στο μηχανισμό χρηματοδότησης. Η Επιτροπή τώρα χρηματοδοτεί βάσει γεωγραφικών προγραμμάτων. Αλλά κάποιες φορές υπάρχουν προγράμματα τα οποία δεν είναι επιλέξιμα για αναπτυξιακή βοήθεια. Το πρόβλημα αυτό επιλήθηκε όταν έγινε δεκτή η έκκλησή μας να προβλεφθεί νέα νομική βάση για τέτοιου είδους μέσα, για την ε, συνεργασία μεταξύ εκβιομηχανισμένων χωρών. Και υπάρχει και μια τεχνικότερη πρόταση. Εδώ η Επιτροπή προτείνει μια πανομοιότυπη ένα πανομοιότυπο μέσο για το μηχανισμό χρηματοδότηση τη αναπτυξιακή συνεργασία και του εκδημοκρατισμού και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για το σκοπό αυτό, εμεί ζητήσαμε να χωριστεί σε δύο ξεχωριστά τμήματα η πρόταση τη ε, Επιτροπή. Γι' αυτό και οι τροπολογίε μα που ζητούν αυτή τη διάκριση μεταξύ του μηχανισμού χρηματοδότηση τη αναπτυξιακή συνεργασία και του μηχανισμού του εκδημοκρατισμού και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και τρίτη μου παρατήρηση, το Κοινοβούλιο θέλει να ασκήσει το δικαίωμα ελέγχου του το 2006 στην τελική φάση των διαπραγματεύσεών μα με το Συμβούλιο και την Επιτροπή για το μηχανισμό αυτό. Συμπεράναμε μετά από δύο, δύο χρόνια δύσκολων διαπραγματεύσεων ότι θα πρέπει να αποδεχτούμε από την αναπτυξιακή προοπτική μια νέα διαδικασία επιτροπολογία που συμφώνησαν μεταξύ του τα θεσμικά όργανα και που αύξησε τι εξουσίε του Κοινοβουλίου. Η ρυθμιστική μεταελέγχου διαδικασία, όπω ονομάστηκε. Ευθύ εξ αρχή φάνηκε ότι για το μηχανισμό αυτό θα πρέπει να εφαρμοστεί ακριβώ αυτή η ε, νέα διαδικασία, καθώ και για τα στατηγικά έγγραφα του μηχανισμού. αλλά η υλοποίηση αυτής της διαδικασίας φαίνεται ότι θέθεται εν κινδύνο τα προγράμματα που περιλαμβάνονται στο μηχανισμό, γι' αυτό δεχτήκαμε την παλιά διαδικασία τροπολογίας. Πολλές φορές αναγκαστήκαμε λοιπόν να δεχτούμε μέτρα, σχέδια μέτρων που πρότεινε η Επιτροπή που δεν συνάδουν με τις διατικές διατάξεις του ίδιου του μηχανισμού χρηματοδότησης. Έτσι, η Επιτροπή υποχρεούται βάσει της νέα διαδικασίας, της διαδικασίας που τώρα ισχύει, να δικαιολογήσει τουλάχιστον ε, την, προ... την πρόταση των μέτρων που κάνει, χωρίς όμως να μπορούμε, μπορούμε να την υποχρεώσουμε να τα αποσύρει ή να τα ανακαλέσει. Πάντω, το Κοινοβούλιο κατά την υλοποίηση του μηχανισμού αυτού ε, επεσήμανε 12 περιπτώσει όπου η Επιτροπή είχε υπερβεί ε, τι προδιαγραφέ που προέβλεπε ο μηχανισμό, ε, δεν είχε σεβαστεί ακριβώ τα κριτήρια επιλεξιμότητα και έτσι αναγκάστηκε να αναθεωρήσει τι προτάσει μέτρων τη και να τι ευθυγραμμίσει με τι ισχύουσε διατάξει. Μόνο σε τρει όμω περιπτώσει η Επιτροπή ανέ, ανέ, ε, ανακάλασε τελείω την πρότασή τη. Το Κοινοβούλιο λοιπόν θα έπρεπε να έχει τη δυνατότητα να μπλοκάρει τελείω τι αποφάσει τη Επιτροπή εφόσον θεωρεί ότι παραβιάζουν τι ε, προδιαγραφέ του μηχανισμού χρηματοδότηση. Η Επιτροπή μα προβλέπει ότι τα στρατηγικά έγγραφα για το μηχανισμό χρηματοδότηση και τα πολιετή προγράμματα θα πρέπει να υπόκεινται στη δικασία επιτροπολογίας ελέγχου και αυτό ζητά το κοινοβούλιο μα συνολικά, Πρόεδρε. Γι' αυτό λοιπόν σε ψήφισμά μα αναφέραμε ρητός από το Σεπτέμβριο του 2008 για την εισαγωγή της ε, νέας αυτής διαδικασίας επιτροπολογίας ελέγχου, ότι θα πρέπει να ισχύει το μηχανισμό αυτό. Η Επιτροπή μάλιστα κλήθηκε να υποβάλει στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο νομοθετική πρόταση για να συμπεριληφθούν εδώ νομικέ πράξει μαζί με το μηχανισμό χρηματοδότηση τη αναπτυξιακή συνεργασία που να υποβάλλονται σε αυτή τη νέα διαδικασία. Η νέα νομοθετική πρόταση τη Επιτροπή για το μηχανισμό χρηματοδότηση δεν περιέλαβε τελικά την ε, διαδικασία αυτή και για αυτό το Κοινοβούλιο ζητά ξανά την υλοποίηση του περσινού του ψηφίσματος. Με την ευκαιρία αυτή απευθύνω έκκληση προς τους συναδέλφους εισηγητές που παρακολουθούν το μηχανισμό χρηματοδότησης και τις εξωτερικές μας δράσεις να ε, συνεχίσουν να ε, συμμετάσχουν στην υλοποίηση όλων αυτών των μέτρων και να ζητήσουν, να επιμείνουν για την εισαγωγή αυτής της νέας διαδικασίας. Πρόεδρο, όπως είπα, τη νέα αυτή διαδικασία επιτροπολογία μεταελέγχου, εφόσον τεθεί σε ισχύ η συνθήκη τη Λισαβόνα, δεν θα καλύπτεται την ίδια νομική βάση, αλλά από το άρθρο 293 της Νέας Συνθήκης. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει τεχνικές δυσκολίες, αλλά αυτά τα επιλύουν οι ειδικοί συνήθως. Γι' αυτό το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή, μαζί με τη Γραμματεία του Συμβουλίου, θα πρέπει να συναντηθούν πριν από τη θέση σε ισχύ τη ε, συνθήκη τη 4 Δεκεμβρίου και θα παραμείνει εδώ στην αρχική μου δήλωση ότι θέλει να αυξήσει τι εξουσίε του το Κοινοβούλιο με την νέα διαδικασία επιτροπολογία και να περάσουμε αυτό το πολιτικό μήνυμα πριν και όχι μετά την 1η Δεκεμβρίου και με την ισχύ των νέων διατάξεων τη συνθήκη. Και αν επιτρέπετε, Πρόεδρε, θα ήθελα να προτείνω να δώσουμε το λόγο στην νομική μα υπηρεσία για να μα εξηγήσει γιατί θα πρέπει να προβλέψουμε την ρυθμιστική αυτή διαδικασία ελέγχου και πώ ακριβώ η αίτησή μα μπορεί να ικανοποιηθεί βάσει των νέων διατάξεων τη συνθήκη τη Λισαμπόνα. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε, λέει πρόεδρο. Να δώσω το λόγο στην νομική υπηρεσία για σχόλια και εξηγήσει. Daniela Gauci from the Λέγομαι Ντανιέλα Γκάουτσι από την νομική υπηρεσία. Ας απαντήσουμε σε ερωτήσεις. Πρώτα, σε ό,τι αφορά την ερώτησή σας για ποιο λόγο θα πρέπει να ζητηθεί η ρυθμιστική διαδικασία με κοινοβουλευτικό έλεγχο, διότι αυτή η διαδικασία ε, εφαρμόζεται όταν ε, πληρούνται τρεις όροι. Τα μέτρα να είναι γενικού χαρακτήρα, τα μέτρα δηλαδή που λαμβάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όταν συμπληρώνουν ή τροποποιούν ε, μια νομοθετική πράξη και όταν έχουν ουσιώδη χαρακτήρα. Τώρα, αντί για την ε, διαχειριστική διαδικασία που εφαρμόζεται τώρα σε έγγραφα στρατηγικής για τα προγράμματα αυτά, η διαφορά είναι ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να προβάλλει δικαίωμα κυρίας απέναντι στις προτάσεις της Επιτροπής. Τώρα, η DCI περιλαμβάνει τα έγγραφα στρατηγικής και ε, προβλέπει ένα συνεκτικό πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ε, περιφερειών, των χωρών δηλαδή, συνεργασίας, με ειδικού στόχους κλπ. Μέτρα τα οποία καθιερώνουν πλαίσια συνεργασιών και ε, τομείς προτεραιοτήτων είναι σαφώς μέτρα γενικού χαρακτήρα. Δεν αναφέρονται δηλαδή σε ένα ειδικό έργο. Στην περίπτωση αυτή άλλωστε συμπληρώνουν αυτά, συμπληρώνουν αυτά που περιλαμβάνονται στο βασικό νομοθέτημα στη DCI. Για το λόγο αυτό λοιπόν υποστηρίζουμε την θέση του εισηγητού. Ότι δηλαδή υπό την ισχύ, ισχύ των ε, ε ισχυσών συνθήκων η ρυθμιστική διαδικασία θα πρέπει να εφαρμοστεί για τα έγγραφα στρατηγική. Σε ό,τι αφορά την ερώτησή σας, πώς μπορεί να αιτιολογηθεί η χρήση αυτής της διαδικασίας υπό τη συνθήκη της Λισαβόνας. Η παρούσα επιτροπολογία, πρώτα-πρώτα, στο άρθρο 202 της παρούσας συνθήκης, Αντί για επιτροπολογία υπό την συνθήκη της Λισαβόνας, θα υπάρχει ένα σύστημα νομοθετικών πράξεων, της ίδιας της DCI δηλαδή, και την δυνατότητα είτε να είναι κατανάθεση, είτε πράξει που εγκρίνει κατά βάση η Επιτροπή. Για τι λεγόμενε την τάξη, αυτέ προσφέρουν περισσότερε εξουσίε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί το 290 άρθρο τη συνθήκη τη Λισαβόνα προβλέπει συγκεκριμένα ότι οι νομοθετικέ πράξει, η DCI εν προκειμένου, περιλαμβάνουν ρητά του όρου υπό του οποίου λειτουργεί η διαδικασία αυτή. Επομένω, αυτοί οι όροι μπορεί να περιλαμβάνουν και το δικαίωμα του Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου να προβάλλει βέτο σε προτάσεις που κάνει η Επιτροπή. Τώρα, σε σχέση με το ποια μέτρα μπορούν να θεωρηθούν κατανάθεση πράξη. πάλι τα κριτήρια είναι γενικής εφαρμογής, συμπλήρωσης ή μη ουσιοδών στοιχείων ε, μιας νομοθετικής πράξης. Άρα παρόμοια κριτήρια με αυτά που έχουμε για την ε, ε, ρυθμιστική διαδικασία με έλεγχο. Όπως εξηγήσαμε, θεωρούμε ότι τα κριτήρια αυτά πληρούνται προκειμένου και γι' αυτό άμα τη θέση ισχύει τη συνθήκη τη Λισαβόνας η αναθεώρηση τη DCI θα πρέπει να λάβει υπόψη και τα έγγραφα στρατηγική και αυτά πρέπει να εγκριθούν ως delegated acts και σε ό,τι αφορά τώρα την ίδια τη διαδικασία επειδή η ψηφοφορία στην Επιτροπή όπως είπατε θα γίνει περί τα τέλη Νοεμβρίου είναι σκόπιμο να παραμείνουν οι τροπολογίες ως έχουν Αναφέρομαι δηλαδή στην ε, ε, ρυθμιστική διαδικασία με ε, κοινοβουλευτικό έλεγχο. Και να γίνουν τα delegate acts πριν από την ψηφοφορία στην Ολομέλεια, αφού αυτά θα μπουν σε ισχύ μετά από τη θέση σε ισχύ τη Συνθήκης Λισαβόνας. Αυτά έχω να πω για την ώρα. Είμαι στη διάθεσή σα για ερωτήσει. Σα ευχαριστώ πολύ. Τα μέλη της Επιτροπή τώρα. Κύριε Ντέβα. Εσείς κύριε Τέβα. Πρώτα πρώτα, συγχαρητήρια για τον συνάδελφο. Επειδή χρόνια δουλέψαμε και είχαμε 16 διαφορετικά νομοθετήματα ε, στα οποία συμμετέσχε το Κοινοβούλιο και μιλούμε για 8 δις ευρώ το οποίο θα κοστίζανε. Και έτσι προσπαθήσαμε να κωδικοποιήσουμε κατά κάποιο τρόπο όλους αυτούς τους κανόνες και να γίνει αποτελεσματική διαχείριση των χρημάτων. Και τότε είχαμε τις εξαιρετικέ αρμοδιότητες της συνθήκης της Λισαβόνας γενικά στο Κοινοβούλιο. Εμεί όμω εδώ στην Επιτροπή Ανάπτυξη χάσαμε αρμοδιότητε. Είχαμε λιγότερε όσον αφορά την εποπτεία του πού πάνε τα χρήματα των φορολογουμένων. Χάσαμε και σε σχέση με την συναπόφαση. Ακούσαμε τη γνώμη των νομικών μα συμβούλων και θα πρέπει να δούμε κατά πόσο μπορούμε να ανακτήσουμε τι αρμοδιότητε για να μπορούμε να παρακολουθούμε και πάλι αυτά που πρέπει. Και αν δεν μπορέσουν να έχουν πραγματικό έλεγχο, τότε δεν διαφέρουν και πάρα πολύ από ένα καφενείο όπου απλώ συζητούμε. Άρα θα πρέπει να δούμε πώς θα δουλέψουμε στο μέλλον. Πώς θα μπορέσουμε να δούμε την αναθεώρηση της ε, συνθήκης Κοτονού και την DCI. Legislative authority. We need to be equally Οπότε να δούμε πως και εμείς θα είμαστε αποφασισμένοι να διατηρήσουμε τις αρμοδιότητες μας ως συνομοθέτες και να μπορούσαμε έτσι να ελέγξουμε την εκτελεστική εξουσία και να μπορέσουμε να ελέγξουμε το πώς δαπανώνται τα χρήματα των φορολογουμένων. Κύριε Μπέρμαν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Συμφωνώ 100% με τον κύριο Ντέβα. Εμεί ακριβώ δίδαμε σε αυτόν τον ρόλο της, του δημοκρατικού ελέγχου. Και θα πρέπει Συμβούλιο και Κομισιόν να καταλάβουν ότι έτσι έχουν τα πράγματα. Η προθεσμία λίγη εξαιρετικά πάρα πολύ σύντομα. Αύριο, αύριο 11, 11 στις 6 ώρα. Εντάξει. Συγγνώμη που αργήσα, αλλά ήμουν σε κάποια άλλη επιτροπή και συζητούσαμε ακριβώ το πράγμα. Δεν μπορούσαμε ταυτόχρονα σε δύο ε, και θέλουμε να δούμε τι θα γίνει με αυτά τα έγγραφα γιατί θεωρούμε ότι θα έχουμε πάρα πολύ σημαντικά προβλήματα εφαρμογή τη συνδίκη και πολιτικά προβλήματα. Ε, θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξουν αυτά τα μέσα πολιτική και έτσι να μπορέσουμε να εκτελέσουμε τον προπολογισμό έγκαιρα του χρόνου. Εκεί είναι το πρόβλημά μας. Με δύο λόγια, αυτή είναι η θέση μας. Ευχαριστώ. Κύριε Μπέρμαν όλοι συμφωνούμε ότι δυστυχώς είναι μια μακρά και δύσκολη διαδικασία η δημοκρατία. Και αυτό το οποίο ο κ. Ντέβα μας είπε τώρα η Επιτροπή είναι απαράδεκτο. Επομένω, θα έχουμε πόλεμο εν συνεχίσει αυτή τη θέση. Πάρα πολύ ξεκάθαρα ε, ε, τοποθετηθήκατε λέει πρόεδρος και οι τροπολογίε θα υποβληθούν και θα προχωρήσουν. Μίτσελ. Ευχαριστούμε τη Γραμματεία και την Νομική Υπηρεσία και τους συναδέλφους για τη βοήθειά τους. Και εμείς θα λάβουμε υπόψη τις νομικές συμβουλές, λέει ο Πρόεδρος. Πάμε τώρα στο επόμενο θέμα μας little shorter. Ε, είναι λίγο συντομότερο. Ανταλλαγή απόψε τον κύριο Πέτερ Τσάγκλ, που είναι ο Γενικό Διευθυντή τη ΕΚΟ, τη Γενική Διεύθυνση για την Ανθρωπιστική Βοήθεια. Είναι εδώ ο κύριο Τζάγκλ. Α, έρχεται, έρχεται.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 Okay. Well, Ξαναρχίζουμε από την αρχή. Συγγνώμη, δεν είδα ότι δεν παρίστασα. Με μεγάλη μας χαρά επομένω, κύριε Τζάγκλ, σας υποδεχόμεθα. Είστε επικεφαλής Γενικό Διευθυντή τη Γενική Διευθύνσεω ΕΚΟ για την Ανθρωπιστική Βοήθεια. Και ξεκίνησατε αυτή την ε, επιχειρησιακή στρατηγική και έτσι έχει τις βασικές προκλήσεις, γεωγραφίες προτεραιότητες, στρατηγικές για την ανθρωπιστική βοήθεια και αρρωγή. Η δε στρατηγική για το 2010 τώρα πρόσφατα προσαρμόστηκε και έχει ηλεκτρονικά διανεμηθεί σε όλους και πολλές από τις χώρες που περιέχονται σε αυτή την ε, ε, στρατηγική κάθε χρόνο ε, αναφέρονται εκεί γιατί έχουμε διάφορες κρίσεις που σοβούν εκεί όπως η Σομαλία και το Κονγκό του χρόνου θα έχουμε δύο αποστολές ερευνητικές στην Παλαιστίνη και στο Νότιο Σουδάν που είναι χώρες ε, που δείχνουν πόσο πολύπλοκη υπόθεση είναι η ανθρωπιστική κρίση. Δε, και του κλίματος, ε, οι ε, όλα αυτά δημιουργούν νέες ανάγκες. Επομένως, και ως ε, αυτά είναι σημαντική η δραστηριότητα της ε, γενικής σας διευθύνσεως. Εμείς θεωρήσαμε ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε και περισσότερο ε, σε αυτές τις ε, δράσεις, όμως θα πρέπει πρώτα-πρώτα να υπενθυμίσω ότι για την ανθρωπιστική βοήθεια έχουμε μια κοινή πολιτική βάση. Την Ευρωπαϊκή Συνένεση για την Ανθρωπιστική Βοήθεια που εγκρίθηκε το 2007. Οι αρχές και οι στόχοι που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα μέλη της χωριστά. Το Κοινοβούλιο από κοντά παρακολουθεί και η Επιτροπή μας επίσης παρακολουθεί την εφαρμογή της ε, στρατηγικής αυτής, της πολιτικής αυτής και έχουμε η Μισελ Στράφερ που είναι αντιπρόεδρος της Επιτροπής και παρακολουθεί συνεχώς ως πάγια, ως μόνιμη ε, εισηγήτρια της ε, εξέλιξης. Κύριε Τζάγκλη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Συγήτρια, κυρίες και κύριοι βουλευτές, επιτρέψτε μου καταρχάς να σας ευχαριστήσω και να εκφράσω τη χαρά μου που για πρώτη φορά στην νέα είμαι στην Επιτροπή σας και με προσκαλέσατε. Ελπίζω ότι η πρώτη αυτή συνάντηση θα αποτελέσει την πρώτη μιας σειράς συναντήσεων συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μια συνεργασία που θα μας επιτρέψει να επικεντρωθούμε στις μεγάλες ανθρωποστικές προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουμε τα επόμενα χρόνια. Να εκφράσω λοιπόν την ικανοποίηση που αισθανθήκαμε όταν δεσμεύτηκε το Κοινοβούλιο και πιο συγκεκριμένα η Επιτροπή ΔΕΒ να συνεργαστεί μαζί μας για τα ζητήματα της ανάπτυξης. Είστε συνεργάτης κλειδί για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσετε να διαδραματίσετε το σημαντικό ρόλο που ως τώρα έχετε διαδραματίσει. Πριν έρθω στις ε, μεγάλες γραμμές της στρατηγικής μας, της επιχειρικής μας στρατηγικής για το 2010, να θυμίσω αυτό που κι εσείς εκφράσατε στα εισαγωγικά σας σχόλια, τη σημασία της συνένεσης για την ανθρωπιστική βοήθεια. Γιατί γιατί ο Επίτροπος όταν του εξήγησα τα περί συνένεσης, μου είπε με την επιφύλαξη των ε, εξελίξεων πρόκειται όλα αυτά είναι ένας κοινός στόχος θα πρέπει να αποτελεί το Ευαγγέλιό μας ε, σε όλη μας τη δράση. Δεν ξέρω αν όλοι συμμεριζόμαστε την ίδια άποψη, αλλά προ αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να κινηθούμε. Και αυτό για μα είναι σημαντικό, γιατί μας επέτρεψε να έχουμε την κοινή έγκριση, τη συνενετική έγκριση των τριών θεσμικών οργάνων για τις τρεις αρχές που διέπουν την υλοποίηση της ανθρωπιστική βοήθεια αρχές που ούτως ή άλλως υπήρχαν, όμως καλύτερα να είναι γραμμένες και σε αποτυπωμένες στο χαρτί και ακόμα και αν επεκτείνονται σε κάποιες σελίδες πέραν του Κοινοβουλίου και των κρατών μελών. Η συνένεση αυτή είναι καρπός μιας διαδικασίας διαβουλεύσεων ε, ευρείας και πλούσιας διαδικασίας που μας επέτρεψε να εξασφαλίσουμε τη συμμετοχή όλων μας των εταίρων. Θα τους αναφέρω αργότερα. Είναι καθοριστική σημασία για την υλοποίηση της βοήθειάς μας και ακόμη και αν δεν είναι επίσημα συμβαλόμενοι στην διαδικασία αυτή, σίγουρα συμφωνούν με τις προτεραιότητές μας. Είναι λοιπόν σημαντικό αυτό και πιστεύω θα το συζητήσετε και αργότερα μέσα στη σημερινή ημέρα. Είναι σημαντικό όλοι μας οι εταίροι να προσυπογράφουν στα σημεία κλειδιά της συνένεσης. Η συνένεση αυτή βασίζεται σε τέσσερις καθοριστικές αρχές. Η αρχή του ανθρωπισμού και εδώ θα θέλω να προσθέσω την αξιοπρέπεια σε μια παρένθεση, η ουδετερότητα, η αμεροληψία και η ανεξαρτησία. Επειδή δεν είμαστε σε ακαδημαϊκό πλαίσιο, βεβαίως δεν θα περάσω σε ορισμούς τώρα, αν θέλετε αργότερα μπορούμε να τα συζητήσουμε και θεωρητικώς. Όπως το έλεγα, το βασικό μας πολιτικό έγγραφο, το πολιτικό έγγραφο αναφοράς, ε, είναι κάτι που θέλουμε να χρησιμοποιηθεί, όχι να μείνει στα χρονοτούλα από των διαφόρων θεσμικών οργάνων. Θα πρέπει λοιπόν τον ενθουσιασμό και το ζήλο μας να τον υλοποιήσουμε. Να φροντίσουμε το consensus, αυτή η συνένεση που έχουμε συντάξει, να χρησιμοποιηθεί με όλο το δυναμικό χαρακτήρα που τον διέπει. Ε, πρέπει να έχει και πολιτική χρήση, αλλά και να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο στις δράσεις μας. Θα πρέπει να μας θυμίζει και ποτέ δεν είναι περιττό να θυμάται κανείς κάποια πράγματα γιατί όταν είμαστε πεπισμένοι για κάτι και έχουμε μια πεποίθηση τίνουμε να ξεχνάμε τις βασικές αρχές πρέπει να σεβόμαστε το διεθνές δίκαιο, το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και το δίκαιο των μεταναστών, των προσφύγων μάλλον. Εδώ τώρα υπάρχει μία σύγχυση ως προς την χαρακτήρα των διαφόρων μέσων. Εδώ δεν έχουμε ένα εργαλείο ακριβώς για την επίλυση των ανθρωπιστικών προβλημάτων. Επιδιώκουμε όμως στόχους ε, βοήθειας, πρόληψης και ανακούφισης από, την, ε, από τον πόνο και τις την αντιμετώπιση των μεγάλων ανθρωπιστικών κρίσεων. Αυτό δεν σημαίνει ότι η ανθρωπιστική βοήθεια δεν θα έχει επιπτώσεις και για τα συστατικά στοιχεία τη διαδικασία διαχείριση κρίσεων, ω προ την πρόληψη ή την διαχείριση κρίσεων. Να σα δώσω ένα παράδειγμα που δεν αφορά μια περιοχή συγκρούσεων με σοβαρά προβλήματα μεν, αλλά θα περάσω αργότερα στο θεωρητικό τμήμα. Στην Κένια έχουμε προγράμματα βοήθειας για την πρόληψη της ξηρασία. Με λίγα λόγια επιτρέπουμε σε πληθυσμού νομαδικού μέσω μιας κεντρικής πολιτικής που βασίζεται στην διαχείριση των υδάτων να αυξήσουν την περίοδο βόσκησης των ε, κοπαθιών τους από τρίμηνο σε έξι με επτά μήνες. Θα γνωρίζετε όλοι ότι η συμβολή στη μείωση των ενδεχόμενων συγκρούσεων με βοσκούς που ζουν στις ε, μεθοριακές περιοχές είναι προφανής. Όσο περισσότερο βόσκηση επιτρέπεται, τόσο λιγότερη σύγκρουση μπορεί να προκύψει. Τόσο λιγότερη ένταση δημιουργείται. Έτσι λοιπόν είναι σημαντικές οι επιπτώσεις, αν και δεν αντιμετωπίζουμε άμεσα την αναχέτηση των ενδεχόμενων συγκρούσεων που μπορεί να ξεσπάσουν. Να λοιπόν ένα είδος παρέμβασης το οποίο μπορούμε να επιχειρήσουμε και το consensus εδώ είναι κάτι που μας καθοδηγεί. Και θα πρέπει και εμείς να ώστε να υπάρχει συνοχή μεταξύ των μέσων απόκρισης της καταστροφές για τις οποίες μπορούμε να έχουμε αρμοδιότητα και τα εργαλεία για τη διαχείριση κρίσεων. Πέρα των βασικών πολιτικών συστατικών του κονσένσους, αυτό το κονσένσους μας επέτρεψε να περάσουμε σε μια θεσμική σημαντική θεσμική αλλαγή, ε, σημαντικό συμπλήρωμα του δικού σας μόνιμου εισηγητή, μόνιμη ομάδα εργασία σε επίπεδο συμβουλίου, το οποίο ονομάζεται, η οποία ονομάζεται ΚΟΑΘΑ, βρισκόμαστε στην εποχή των συντομογραφιών και ασχολείται με την ανθρωπιστική βοήθεια και την ε, ανάπτυξη. Τα τελευταία τρία χρόνια ασχολείται όχι μόνο λοιπόν με το σκέλο τη ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά με την επισητιστική πιο συγκεκριμένα. Οπότε η ομάδα αυτή εργασία ανταποκρίνεται ακριβώ στην εντολή που έχουμε αναλάβει. Μα επιτρέπει λοιπόν η ομάδα αυτή να επιβλέπουμε την υλοποίηση τη ανθρωπιστική διάσταση κατά τη διαδικασία λήψη αποφάσεων. Και αυτό στο επίπεδο του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων. Η ομάδα ξεκίνησε τις εργασίες τη την 1η Ιανουαρίου και για την ώρα είμαστε ικανοποιημένοι με την πρόοδο που έχει επιτελέσει. Πέραν αυτών, το κονσένσου μα καθοδηγεί όταν προσπαθούμε να ορίσουμε και οριζόντιε προτεραιότητε, στι οποίε αφιερώνουμε και πόρου από τον προπολογισμό. Και βεβαίω να καταρτήσουμε καλύτερα την επιχειρησιακή μα στρατηγική. Σε αυτό το πλαίσιο τη στρατηγική μα θα σημειώσω ότι υπάρχουν τρία βασικά σχόλια που πρέπει να γίνουν αλλά για τα οποία δεν έχουμε ακριβώς εμείς τον έλεγχο. Πρώτον, η αύξηση του ευάλωτου, του χαρακτήρα του ευάλωτου που έχει να κάνει με τους μεταποτιστέντες, τους πρόσφυγες, μετά από ένοπλες συγκρούσεις όπως έγινε στο Πακιστάν, τη Σριλάνκα, τη Σομαλία. Ξέρετε ότι ο κατάλογος είναι μακροσκελής. Δε χρειάζεται να αναφέρω άλλες πέραν από τις πιο των πιο πρόσφατων κρίσεων. Ένα δεύτερο στοιχείο που καθορίζει την προτεραιότητα παρέμβασή μα είναι η αύξηση των φυσικών καταστροφών που συνδέεται ω προ τον αριθμό μάλλον και τι επιπτώσει που έχουν προκύψει από τι κλιματικέ αλλαγέ. Τρίτο στοιχείο, οι τιμέ. Η έκρηξη των ε, τιμών των τροφίμων το 2008. Ακόμα και αν ε, μετριάστηκαν κάπως οι τιμές σε παγκόσμιο επίπεδο, η διάθεση προϊόντων στις ζώνες παρέμβασης δεν έπαψε. Τα συζητήσατε νομίζω χθες, προβλεπόταν το σημείο αυτό στην ημερήσια διαταξή σας. Το φαινόμενο αυτό λοιπόν έκρηξη των τιμών διωγγώθηκε από την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση. Οπότε ο αριθμός των ατόμων που βρίσκονται σε κατάσταση υποσυτισμού και πρέπει να βοηθηθούν και να στηριχθούν φτάνουν, αγγίζουν πλέον το 1 δις, ε, δισεκατομμύριο. Ο αντίκτυπο βεβαίω ε, διωγγώνεται λόγω της ε, χρηματοπιστωτικής και οικονομική κρίση, όπω ήδη το είπα. Οι αυξημένε αυτέ ανάγκε που προκύπτουν από αυτά τα τρία περιοριστικά στοιχεία περιλαμβάνονται σε ένα δυσχερέ πλαίσιο των ε, φραγμών, των δυσκολιών του προπολογισμού που όλο ένα και αυτά διωγγώνονται. Το γνωρίζει το Κοινοβούλιο, υπάρχουν περιορισμοί στον δημοσιονομική, δεν θα επεκταθώ σε αυτό. Αλλά πριν περάσω στην συνέχεια, μάλλον πριν προσπαθήσουμε να χρησιμοποιήσουμε περισσότερους δημοσιονομικούς πόρους, να θυμίσω ένα έγγραφο που έχουμε μοιράσει εδώ. Θα δείτε εκεί ότι η αύξηση των δημοσιονομικών πόρων που αποδίδονται στην Γενική Διεύθυνση ΕΚΟ από το 2007-2010 ε, αυξήθηκαν κατά 30 εκατομμύρια ευρώ. Λιγότερο από 5%. Μην σχολιάσω τώρα, νομίζω ότι η αριθμή είναι εύκολη. Πρόκειται για το πλαίσιο που αποτελεί την πραγματικότητά μα. Εντό αυτού πρέπει να λειτουργήσουμε. Σα το λέω απλώ ενημερωτικά. Για το τι συμβαίνει τώρα στην πράξη. Τρία παραδείγματα συγκεκριμένων προβλημάτων που δείχνουν ότι αυξάνεται η ανάγκη για ανθρωπιστική βοήθεια και ότι πρέπει να αυξηθεί και η δυνατότητα παρέμβασής μας στις ε, ζώνες με πάρα πολλέ δυσκολίε. Δηλαδή λιγότερες ποσότητες με αυξημένες τιμές. Να τι εμπόδια πρέπει κανείς να υπερβεί για να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες αλλά να καλύψει και το απαιτούμενο κόστος. Γνωρίζουμε λοιπόν ότι έχουμε τις, ε, τους ε, καταναγκαστικούς εκτοπισμούς, ε, σεξουαλική βία κατά των παιδιών και των γυναικών, σημαντική διάσταση αυτή για τα παιδιά και τρίτον η στρατολόγηση σε παιδική ηλικία. Να μερικά παραδείγματα. Πέραν αυτών των πρόδειλων και τακτικών παραβιάσεων, οι απειλές ε, κατά του ανθρωπιστικού πλαισίου αυξάνονται. Εδώ, χωρίς τους ανθρωπιστικούς μας εταίρους, δεν θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε να χορηγούμε βοήθεια, κάτι που θα ήταν δραματικό. Σε πολλές περιπτώσεις ε, το ανθρωπιστικό πλαίσιο συρρυκνώνεται, γιατί μας, ε, γίνεται, μας αρνούνται την πρόσβαση τα πράγματα είναι πολλές φορές πολύ δύσκολα, όπως ε, στη Βρυμανία πριν ε, από ένα χρόνο ή στη Σρι Λάνκα πρόσφατα. Βλέπουμε, βέβαια να μας λένε οι πρόσφατες πληροφορίες ότι η κατάσταση στη Σρι Λάνκα βελτιώνεται, αλλά σήμερα στο Πακιστάν η, πρόσφαση, η πρόσβαση στις ζώνες όπου πρέπει να παρέμβουμε είναι δύσκολη. Δεν υπάρχει καν εξουσιοδότηση και ούτε για τους ε, υπόλοιπους διεθνείς φορείς ανθρωπιστικής βοήθειας υπάρχει τέτοια πρόσβαση. Έπειτα, ο συνδυασμός των ρόλων μας είναι κάτι που θα χρειαστεί να προβλέψουμε στο μέλλον. Δύο είναι οι φορείς που συχνά βλέπουμε να κυκλοφορούν με ένα ανθρωπιστικό λογότυπο. Είναι συχνά στρατιωτικής προέλευσης. Δεν κριτικάρα τώρα τους στατιώτες και τους στρατιωτικούς. Πολλές φορές έχουν και πολιτική εντολή, εντολή πολιτικού χαρακτήρα. Αλλά τους δίδεται συχνά μια ψευδοεντολή Δηλαδή από... Ε, δεν είναι το ίδιο ένα σάκος ε, με τρόφιμα που δίνεται από ένα στρατιώτη και από μια ανεξάρτητη ανθρωπιστική αποστολή. Πρέπει λοιπόν να έχει κανείς υπόψη να πρόκειται για παράγοντα ανθρωπιστικής αποστολής ή στρατιώτη. Και βεβαίως αυτό μας φέρνει και στην προστασία των πολιτών, σημαντικό για την προσέγγιση των πολιτισμών στην πράξη βλέπουμε να λειτουργεί σωστά η διαδικασία αυτή. Δεν έχουμε ξυπνήσει κανένα πρωί με ξαφνικές εκπλήξεις. Αλλά δεν θα έλεγε κανείς ότι η προσέγγιση μας έχει καταλήξει στο να περπατάμε και χέρι-χέρι με τους ε, πληθυσμούς ε, που βοηθάμε. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πιο ενεργοί και στη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων ε, παραγόντων, ε, στη συνεργασία με τις ιδιωτικέ εταιρείε, τις μη οργανώσεις και το καθεξής. Τώρα πιο συγκεκριμένα η στατηγική μας, οριζόντια στοιχεία και στοιχεία γεωγραφικά. Στα οριζόντια στοιχεία έχουμε την απόκριση στις επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών με μια ανάμειξη προγραμμάτων προετοιμασίας για τους κινδύνους και τις δυνατότητες απόκρισης. Έδωσα προηγουμένως κάποια παραδείγματα. Προγράμματα για την κένια προετοιμασίας έναντι της ξηρασίας και τα προγράμματα Ήπικο για την προετοιμασία αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών στο Μπαγκλαντές, στο Βιετνάμ και στην καυτή επικαιρότητα στο Ελ Σαλβαντόρ όπου τέσσερις επαρχίες εφαρμόζουν τέτοια προγράμματα επεκό. Χθες μάλιστα και προχθές αυτή η προετοιμασία τους τους επέτρεψε να μετακινήσουν πληθυσμούς σε διαμερίσματα που επλήγησαν από τον ε, πρόσφατο κυκλώνα. Τα μέτρα λοιπόν αυτά προετοιμασίας πολλές φορές μεταφράζονται από χειροπιαστά αποτελέσματα που ακόμα και αν δεν έχουμε αξιόπιστη ροή πληροφοριών, δείχνουν ότι ένα αυξημένο αριθμό του ντόπιου πληθυσμού έχει μπορέσει να προστατευτεί από τι ε, απειλέ των φυσικών καταστροφών. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ πολύ σύντομα και στην ε, δημοσίευση που κάνουμε σε τακτή χρονική βάση στον, στο τοπό μας κάποιων εγγράφων. Έφερα μαζί μου κάποια αντίγραφα των ε, πρακτικών του ιστότοπου για την περίπτωση του Ελσαλβαντόρ. Επιτρέψτε μου αυτή τη διαφημιστική κίνηση. Σας τα έφερα τα έγγραφα αυτά για να δείτε ότι παρακολουθούμε τις εξελίξεις από πολύ κοντά και είναι και έγγραφα τα οποία μπορείτε να τα δείτε και για της ηλεκτρονικής οδού. Επειδή οπτικός όμως μπορεί να μην έχετε εικόνα των εγγράφων αυτών, θεώρησα ότι και οπτικός αλλά και για την αφή είναι σημαντικό να τα δείτε και εδώ μπροστά σας σήμερα. Γι' αυτό σας τα έφερα στην αίθουσα. Το δεύτερο οριζόντιο στοιχείο είναι η έρευνα, η εντατική έρευνα για την επισητιστική βοήθεια. Ε, ιδιαίτερο σκέλος της ανθρωπιστικής βοήθειας ως προς την ανάπτυξη. Νομίζω εδώ είναι σημαντική η τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη της βοήθειας. Δηλαδή να ξεκινήσουμε από μια παλιότερη έννοια. Να φορτώνουμε λόγω χάρη καράβια με εντυπωσιακού όγκους τροφίμων. Ε, αυτό είναι μια παλιά αντίληψη. Στο να περάσουμε στην τόπια παραγωγή των τροφίμων. Αυτή είναι η νέα, η σύγχρονη προσέγγιση. Το τρίτο στοιχείο είναι η προστασία του κοινοτικού, με συγχωρείτε, του ανθρωπιστικού χώρου. Επιτρέψτε μου επίσης ε, σε αυτό το πλαίσιο να θυμίσω το λογότυπο LLD Link Relief Recovery σημαίνει στα αγγλικά Πρέπει να κάνουμε εδώ ό,τι μπορούμε και βάσει αυτό το λογότυπο. Θα πρέπει να το στηρίξουμε περαιτέρω και επειδή μου δώσατε 15 λεπτά πρόεδρε και τα έχω σχεδόν εξαντλήσει δώστε μου ακόμη δύο για τις γεωγραφικές μας προτεραιότητες. Οι γεωγραφικές μας προτεραιότητες υπαγορεύονται από το που υπάρχουν ζώνες συγκρούσεων. Ουσιαστικά μιλάμε για την υποσαχάρια Αφρική για το 2010 για το Σουδάν, το Τσάντ, το κέρας της Αφρικής με τα προβλήματα της ξηρασίας που είναι πολύ σοβαρά και την Κεντρική Αφρική σας είπα περίπου τι προβλέπουμε έχουμε ένα ποσό που ξεπερνά τα 280 εκατομμύρια έχουμε στη θέση μας 800 περίπου εκατομμύρια προγραμματίσαμε ήδη τα 620 και έχουμε Τέσσερι ζώνες υπόψη να καλύψουμε με αυτά τα κονδύλια, πάνω από τέσσερι ζώνες. Μιλάμε εδώ για κατεχόμενα εδάφη, τα κατεχόμενα της Παλαιστίνης, που όμως δεν θα καλυφθούν και το 2010 με τον ίδιο τρόπο. Αμέσως μετά έρχονται το Πακιστάν και το Αφγανιστάν, που το 2009 ε, καλύψαμε με 100 εκατομμύρια ευρώ προβλέψαμε το 2010 πολύ λιγότερα για το Πακιστάν για δύο λόγους. Γιατί ένα μέρος της βοήθειας που αποφασίστηκε το 2009 δεν θα εκτελεστεί το 2010. Δεν μπορεί να υπάρχει διαρκής βοήθεια και επειδή υπάρχει και αυτό που έλεγα προηγουμένως, ότι πρέπει πρώτα να βεβαιωθούμε ότι μπορούμε να διαθέσουμε τα κονδύλια, τη βοήθεια, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων Δηλαδή οι εταίροι μας να μπορούν να λάβουν και να διανύμουν τη βοήθεια. Είμαι πολύ αυστηρός αυτό και το θεωρώ πολύ σημαντικό στοιχείο. Δύο ακόμη αριθμοί για τα προγράμματα παρέμβασης. Εδώ καταβάλουμε ιδιαίτερες προσπάθειες από το 2009 προς το 2010. Όλα τα προγράμματα προετοιμασίας για την πρόληψη, το 2009 κόστησαν γύρω στα 40 εκατομμύρια, Τώρα προβλέπουμε να διαθέσουμε 75 εκατομμύρια για να καλύψουμε αυτή τη διάσταση. Και είναι λογικό αυτό γιατί ένα ευρώ επένδυσης για προετοιμασία αποδίδει πολύ περισσότερα από ότι ένα ευρώ που επενδύεται τη στιγμή της κρίσης. Τελευταία παρατήρηση, πραγματικά ακροτελεύτια, η σημασία των κρίσεων. Θα βρείτε τον κατάλογο στο έγγραφο που σας μοιράστηκε επικεντρωνόμαστε σε 12 από τις κρίσεις που έχουν ξεχαστεί. Να σας θυμίσω τις δύο πιο χαρακτηριστικές για να έχετε υπόψη γιατί μιλάμε. Για την Κολομβία, όπου χρόνο, με το χρόνο παρά τη βελτίωση της στατιωτικής κατάστασης, μεν έχουμε 300.000 εκτοπιστέντες στο εσωτερικό της χώρας. Ε, ε του συνδράμουν οι Κολομβιανέ αρχέ του ανθρώπου αυτού, αλλά όχι αρκετά. Υπάρχουν διάφορες ε, ε, εθνότητες εδώ που καλύπτονται, αλλά η Σάουαουι είναι πιο χαρακτηριστική, αλλά υπάρχουν κι άλλε καμιά δεκαριά. Και τελευταία παρατήρηση, θεσμική, επιτρέψτε μου τελευταία πρόταση, Πρόεδρε, το δικαίωμα ελέγχου του Κοινοβουλίου. Να σας ευχαριστήσω εδώ για το επικοδημοτικό πνεύμα της συνεργασίας μας και την ε, ταχύτητα με την οποία εξετάζετε τα θέματα τα οποία μας επιτρέπουν να καλύπτουμε τις προθεσμίες, να ανατηρούμε τις προθεσμίες και βεβαίω ε, δίνεται και την σημασία που αρμόζει στις παρεμβάσει μα. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, με στη διάθεσή σα. κύριε και τώρα. Ε, θα, έχει πάγια, μόνιμη, διαρκής συγκεκριτικά μας κύριε Στυβλέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω κάποιε παρατηρήσει και κάποιε ερωτήσει από αυτή τη στρατηγική πρώτα όσον αφορά αυτή την κρίση του Σαχέλ. Εδώ Τσάντ, Μαλή, Μαυρετανία, ε, Νίγηρα. Ε, είναι μια κρίση σχεδόν ε, ξεχασμένη γιατί εκεί έχουμε εξωτερικού παράγοντε όπω πολιτική αστάθεια, απερίμωση και άλλους που παραξύνουν μια κατάσταση που ήδη είναι κακή, χωρίς όμως να μπορούν να τραβήξουν την προσοχή των ΜΜΕ. Πήγα στην να φάσω πρόσφατα στα πλαίσια της ε, συνάντησης της περιφερειακής της ε, ΑΚΕ και θα πρέπει να ευχαριστήσω άλλη μια φορά την ΕΚΟ και τους ε, επιτόπου υπαλλήλους γιατί οργάνωσαν αυτή την αποστολή την επιστολή μετά από τις πλημμύρες αυτές στην Ογκαντούγκου και συναντήσαμε τοπικού παράγοντε. είδαμε τι, μπορεί, τι, κάνει για όλο αυτό το τον κόσμο ε, η ΕΚΟ. Τώρα να δούμε τι χρηματοδοτικά μέσα μπορούμε να επιστρατεύσουμε το 2010. Τι μπορεί να προοικοδοτηθεί το 2010 ούτω ώστε αυτή τη διατροφική κρίση του Σαχέλ να την αντιμετωπίσουμε. Ε, Επίση να ε, πέσει η θνησιμότητα, σταματήσει η κακή διατροφή όλων αυτών που βρίσκονται σε τόσο επικίνδυνη, δύσκολη θέση. Το 2009 δόθηκε επιπλέον βοήθεια, 8 εκατομμύρια ευρώ, το ώστε να καταπολεμηθεί η ξηρασία της Κένιας. Επίσης, είχαμε πει ότι θα πρέπει μια δική μας ε, αντιπροσωπεία να μεταβεί στην περιοχή του 2010. Θα πρέπει να ζητηθεί με ποια μέσα η ΕΚΟ μπορεί κάτι να κάνει για αυτή την κρίση. Όσον αφορά Κάποιε θεομηνίε το 2010 μπορεί η Κομισιόν να απευθυνθεί στι αρχές του προπολογισμού τόσο ώστε από το ειδικό κονδύλιο να εκταμιεύσει κάποια χρήματα ε, πέραν της ε, ανθρωπιστικής βοήθειας. Εσείς θεωρείτε ότι αυτή η επίγουσα βοήθεια του 2010 θα αρκέσει και τι ποσό από αυτήν την έξτρα επίγουσα βοήθεια χρησιμοποιεί το 2009 επίσης λόγω αυτών των περιορισμών της κυβέρνησης για πέστε μας υπάρχει προγραμματισμός όσον αφορά ε, το τι θα κάνετε το 2010. Το 2009 δεν υπήρξε. Τώρα, όσον αφορά την διεθνή ανθρωπιστική βοήθεια, τι μπορεί να γίνει για να αντιμετωπίσει αυτή η κατάσταση. Επίσης, δεν έχετε προσυπογράψει την συνθήκη της Γενέβης. Βεβαίως όμως βοηθάτε όσον αφορά την διανομή της διεθνού βοήθειας. Πεςτε μας τι δράσεις της Κομισιόν το 2010 μπορεί να γίνουν ούτω ώστε να συνεχιστεί αυτό το πλαίσιο και να μπορεί να υπάρχει προσβασιμότητα των ε, πλέον ευάλωτων ε, στην ανθρωπιστική βοήθεια. Τώρα, όσον αφορά τη συνθήκη της Λισαβόνας, κλείνω, κλείνω. Με συνθήκη της Λισαβόνας ε, πρέπει να δούμε ότι θα υπάρξει νομική βάση το, το άρθρο 114. Θα έχουμε δε την υπηρεσία για εξωτερική δράση. Επομένως, ποιες θα είναι για την ΕΚΟ οι συνέπειες, τι αυτονομία δράσης θα έχει η ανθρωπιστική βοήθεια. Προβλέπεται στο πρόγραμμα δράσης η Κομισιόν του 2010 να κάνει μια ενδιάμεση αναθεώρηση, ούτως ώστε να δούμε τι θα γίνει με την συνένεση με τους εταίρους μας. Οπότε μπορείτε μήπως να μας ενημερώσετε από αυτού να δούμε τι οργάνωση υπάρχει και τι διαδικασία προβλέπεται. Τώρα, αν θα υπάρξει ε, έκθεση δίας πρωτοβουλίας, δεν ξέρω. Η πρόεδρος. Καλά. Ε, κ. Κάσμαρκ τώρα έχει τον λόγο στα πολωνικά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Διευθυντά, ευσύνοπτη η προσοχή και ευχαριστούμε. Για την Ερυθρέα προβλέπονται απεσιόδοξα πράγματα, απεσιόδοξε εξελίξεις. Τίποτα δεν έχει ε, προβληθεί. Δύσκολα είναι και τα πράγματα. Υπάρχουν προβλήματα διατροφή κλπ. Όμω, για στρατηγικούς λόγους, νομίζω, θα μπορούσαμε να προσδοκούμε κάποια βήματα προόδου. Όπως νερό για τους ποιμένες. Και μπορεί να γίνουν κάποια μακρόπνοα ε, προγράμματα. Τι μπορούμε να κάνουμε για την Ερυθρέα, για πετε μας. Υπάρχει τελικά ελπίδα το 2010 να έχουμε κάποια προγράμματα, κάποια έργα Φερρυπίν, ανέγερση φραγμάτων. Κάτι να γίνει για την ίδρυυση της χώρας. Ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος, και δίνω το λόγο στον κύριο Γκερέρο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε, κύριε Γενικέ, για την εισήγησή σας. Θεωρώ ότι η ανθρωπιστική βοήθεια είναι μια ένδειξη. Ένδειξη του ηθικού μεγέθους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε όσο πιο σημαντική είναι αυτή η ανθρωπιστική βοήθεια, όσο περισσότερο ανταποκρινόμαστε στη Σολένα και περισσότερες ανάγκες που ανακύπτουν, τόσο περισσότερο θα αναγνωρίζεται η ηθική μας πλευρά. Τώρα, να επισημάνω κάτι το οποίο φαίνεται περιθωριακή σημασία, μικρή σημασία, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό για την νόμη. Δηλαδή το ότι θα πρέπει κάτι να κάνουμε ούτω ώστε να εξασφαλίσουμε την, την, ασφάλεια, του εύρυθμου όρου λειτουργία όσων βοηθούν για την ανθρωπιστική βοήθεια. Γιατί το έργο του είναι δύσκολο. Είναι μια θυσία. Όμω βλέπουμε ότι του τελευταίου μήνε ρισκάρισαν την ίδια τη ζωή του. Και δεν είναι τελικά θέμα δικαιοσύνη. Είναι θέμα και αποτελεσματικότητας Τη ίδια μας ανθρωπικής βοήθειας. Διότι αν δεν υπάρχει ασφάλεια στους όρου που επιτελούν το έργο τους τότε δεν θα μπορέσουν να επιτελέσουν το έργο τους και να βοηθήσουν αυτού που χρειάζονται την ανάγκη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Γενικό για τα όσα μας είπε όσον αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια. Έχω να σας ρωτήσω κάτι. το κλιματικό πρόβλημα. Πώς ε, θεωρείτε ότι συμβαδίζει με την ανθρωπιστική βοήθεια στην Κένια ας πούμε. Γιατί υπάρχει εκεί πέρα το πρόβλημα των βοσκοτόπων. Έχουμε τα θέματα της ε, αναδάσωσης, αυτό το Green Belt Movement. 30 εκατομμύρια φυτά έχουν ε, φυτευτεί. Και ξέρετε, τελικά εκεί έχουμε ε, υπερβολικό, υπερβολική βόσκηση. Επομένως, έτσι έρχεται η απερίμωση και δυσκολεύεται μετά βέβαια η ανθρωπιστική βοήθεια, δυσκολεύεται η κατάσταση εκεί και άρα μπαίνουμε σε κάποιο φαύλο κύκλο. Τι μπορούμε να κάνουμε εκεί και τι γίνεται με την κλίμα, του Γκέρεντς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα όσα χρήσιμα μας είπε ο κύριος Γενικός. Τώρα θέλω να σταθώ σε αυτό που ονομάσατε αμάλγαμα. Για την ψυχή βοήθεια την ένστολη και την χωρίστολη. Χρειάζεται να υπάρχει συνέπεια στις πολιτικές μας. Όταν κανείς ενεργεί για την ανθρωπιστική πολιτική της ΕΕ, όμως όταν παράλληλα ασκεί και στρατηγικές επιχειρήσεις ΕΕ, τότε τι γίνεται με το περίφημο αμάλγαμα, Άλλη ερώτηση. Μας ανησυχεί πάρα πολύ το πόσο κινδυνεύουν οι άνθρωποι που δουλεύουν για την ανθρωπιστική βοήθεια, ιδίω στην Ανατολική Αφρική. Που κινδυνεύουν εκεί από τους τρομοκράτες που δρούν στην περιοχή εκείνη. Μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια παραπάνω όσον αφορά το τι γίνεται εκεί, τη διακινδύνευση που υπάρχει. Η πρόεδρος. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω να ζητεί άλλο το λόγο. Οπότε, θα δώσω ξανά το λόγο στον κύριο Ζάγκελ. Πολύ με... μακρύς αυτός ο κατάλογος. Όμως θα αρχίσω από την ερώτηση της κυρίας Στρίφλα. Μας είπε για την να φάσω όπου είχε πάει, ήταν πάρα πολύ σαφές το μήνυμα για μας. Έγινε το πρώτο βήμα. Είναι απλά το πρώτο βήμα, που θα συνεχίσετε προς αυτήν την κατεύθυνση και είναι πολύ σημαντικό, γιατί τίποτα δεν μπορεί να την καταστήσει το να πάει κανείς επιτόπου για να δει την κατάσταση. Με τη σειρά θα σας απαντήσω, αλλά επ' αυτού. Είπατε για το κατεπήγον, όμως η ανθρωπιστική βοήθεια δεν έχει πάντα κατεπήγοντα χαρακτήρα. Θα πρέπει κανείς να προστατευτεί από αυτή την αντίδραση. Δεν είναι όλα τις κατεπηγούσεις αντίδρασης και γι' αυτό και έχουμε προγραμματισμό. Προσοχή, είπαμε ότι ε, κινδυνεύουν να απορροφήσουν το 80% των κονδυλίων του 2010. Προσοχή γιατί υπάρχει ανάγκη. Αυτά. Όσον αφορά τώρα τη συγκεκριμένη ερώτηση για το Σαχέλ. Για το 2010 έχουν προβλεφθεί 20 εκατομμύρια. Υπάρχει αυτό το περιφερειακό πρόγραμμα για την ε, ξηρασία, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το λέμε και το ξαναλέμε γιατί έχω ασχοληθεί και σε άλλες υπηρεσίες της Κομισιόν και πάρα πολύ σημαντικά ποσά διατίθενται για το ίδιο πρόβλημα που είναι ποσά πολύ πιο μεγάλα. Ε, για την, για την ανθρωπιστική υπηρεσία τα 20 εκατομμύρια είναι πάρα πολλά. Μισό εκατομμύριο να πάει σε μία και μόνη χώρα σαν πίστοση αυτό θεωρείται φανταστικό. Άρα 20 εκατομμύρια είναι πολλά για μας σε σχέση με το σύνολο των παρεμβάσεων που κάνουμε τώρα. Επίση, μα είπατε τι γίνεται με αυτό το υποθεματικό τη κατεπηγούση ανάγκη και το υποθεματικό αυτό ευτυχώ που υπάρχει. Και το χρησιμοποιούμε σταθερά κάθε χρόνο. Έγινε μία μόνο εξαίρεση σε μία δεκαετία. Το δε 2009 εκταμιεύτηκαν 110 εκατομμύρια παραπάνω από αυτό το αποθεματικό για την ξηρασία. Για το κέρας Αφρικής ε, θεωρητικά πήγανε, αντί για το Σαχέλα, εν πάση τόση όμως αυτά χρησιμοποίησαμε. Και έτσι μπορέσαμε να χρηματοδοτήσουμε και κάποιες ευξημένες ανάγκες του Πακιστάν. Το πρόβλημα υπάρχει. Το έχετε και εσείς, το έχουμε και εμείς και συζητήθηκε στο Συμβούλιο. Το μήνυμά σας επομένως ε, το λάβαμε. Τώρα, όσον αφορά αυτό το ερώτημα που έχετε θέσει, δηλαδή το πώς θα μπορέσουμε να δράσουμε υπάρχει κάτι που δεν σας είπα. 122 συνεργάτες μας σκοτώθηκαν το 2008 ενώ εκτός των καθηκοντών τους κάτι το οποίο είναι κάτι το οποίο είναι μεγαλύτερος νούμερο από το πόσοι σκοτώθηκαν από την ειρηνευτική δύναμη. Επομένως, η ανησυχία είναι πάρα πολύ σοβαρή. Στις 31 Δεκάτου ΔΕΠ, που θα να κάνουμε τον απολύσμα του 2009 θα έχουμε περισσότερους νεκρούς που θα έχουμε καταμετρήσει. Και εγώ κάθομαι και συντάζω αυτές τις επιστολές συλληπιτηρίων που αφορά τα θύματα των διαφόρων φορέων που συνεργάζονται για την ε, ανθρωπιστική βοήθεια. Εμείς είμαστε απλώς ένας εκ των πολλών. Επομένως, η κατάσταση είναι πάρα πολύ ενισχυτική. Και δεν φαίνεται να βελτιώνεται. και μην ε, θεωρείτε ότι η απάντηση είναι πολιτικός διάλογος σε ανώτερο επίπεδο. Πρέπει να προσπαθήσουμε σε όλα τα επίπεδα, σε τοπικό, σε ανώτατο, σε ενδιάμεσο, με όλους τους εμπλεκόμενους. Και υπάρχουν Πολλοί λόγοι του οποίου πρέπει να φοβάται κάποιο συνεργάτε μα. Τα όπλα. Τα ξέρετε. Τα τεθωρακισμένα αυτοκίνητα. Οπότε τελικά χρειάζεται και η πρακτική προστασία. Και ζουν σε προστατευμένο περιβάλλον. ας πούμε στο Πακιστάν δεν μένουν σε ξενοδοχεία, μένουν σε ειδικά φυλασσόμενα μέρη. Και πρέπει επίσης να υπάρχει συνομιλία με την πραγματική εξουσία τους τοπικούς παράγοντες. Όλοι αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική για την ασφαλεία μας. Βέβαια, καταλαβαίνετε, με 122 νεκρούς δεν και τα πράγματα τόσο τέλεια. Από την άλλη μεριά όμως, με τα παραδοσιακά μέσα όπως η συνοδεία, τεθωρακισμένα όπως είπατε κι εσείς για την ανθρωπιστική βοήθεια, την ένστολη και την μία ένστολη υπάρχει εδώ πέρα ένα πρόβλημα όμως που δημιουργεί διότι θα πρέπει οι αποδέκτες της βοήθειας να γνωρίζουν τι είδους βοήθεια λαμβάνουν Εδώ είναι τώρα το θέμα της εξαρτησίας, της ουδετερότητας. γιατί θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τι συνέπειε τη βοήθειάς μας όσον αφορά την επίλυση του προβλήματο, γιατί πεθαίνουν από την πείνα, δεν έχουν σπίτι οπότε τι διάλογο να, να, να γίνει με αυτού του ανθρώπου όσον αφορά τι ε, προοπτικές της κατάστασης όμως όταν έχει να αρχίσει να καλύπτει το διατροφικό πρόβλημα ή το στεγαστικό τότε μπορεί να ξεκινήσει ο διάλογο για επίλυση της κρίσης. Σα τα λέω για να καταλάβετε πώ σκέφτομαι. Κάτι άλλο το οποίο το είπε και Στίφλερ που πήγε επί τόπο Ναι, προβλήθηκε εκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρουσία Οπότε και εμείς έτσι ενεργούμε. Δεν, δεν κρυβόμαστε ποιοι είμαστε. Το αντίθετο. Και πολλές φορές οι εταίροι μας δυσφορούν. Προσπαθούμε λοιπόν να δείξουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εκεί και βοηθάει. Επομένως, αυτή, υπάρχει μια διεκτική σχέση μεταξύ ανεξάρτητης ενέργειας και προβολής. Ενδιαφέρουσα αυτή η διαλυτική σχέση. Έτσι βλέπετε λοιπόν, δεν, δεν πατάμε το κουμπί σε ένα υπολογιστή και να πούμε να έτσι διατίθεται αυτά τα χρήματα. Στην Πουρκίνα το είδατε κύριε Στίφλερ. Έχουμε εκεί πέρα κάποιου εμπειρογνώμονε, κάποιου επαγγελματίε οι οποίοι πήγαν εκεί, κάποιοι άλλοι πήγαν στο Σαλβαδόρ και πρώτα ε, πρώτα πηγαίνουν, καταγράφουν παντού ποια είναι τα προβλήματα, θεομηνίε, οτιδήποτε. Ε, οπότε και έτσι έχουμε μια βάση υπολογισμού και έτσι υπολογίζουμε αντί για το κουμπάκι του υπολογιστή το ποσό που χρειάζεται. Να και με τη δυνατότητα βέβαια. Άλλα κάνουμε στην Αιτία, άλλα κάνουμε στο Λοδόρ βέβαια. Όμω, πάντα ενεργούμε εξάρτητα. Δεν ζητάμε κανό είδου συνδρομή από κάποια αρχή για να μας πει πόσα θα χρειάζονται. Πάντοτε έχουμε διάλογο, πάντοτε του ενημερώνουμε, Όμω, δεν ζητούμε ποτέ κανό είδου διαπραγμάτευση, έγκριση από τις αρχές για το ποσό το οποίο ενδεχομένω χρειάζεται. Βεβαίω και ακούμε τι λένε, γιατί θα είναι χαζό να μην ακούμε κάποια τοπική αρχή που ξέρει. Φτάσαμε αυτό το ανθρωπιστικό, είναι θέμα το οποίο ανακύπτει συνεχώς. Γιατί πολλές φορές ζητούμε βοήθεια. Πολλές φορές ζητείται απλά και μόνο η ειδική βοήθεια, ας πούμε για το Νταρφούρ που τόσο συχνά ανακύπτει και θα, το, θα, το, ξαναβγεί το θέμα για το Σουδάν. Για τη Λισαβόνα, το συνήθι της Το μεγάλο πλέον έκτημα είναι ότι η ανθρωπιστική βοήθεια θα προβλέπεται ως αυτόνομη πολιτική κοινή αρμοδιότητα. Συναρμοδιότητα, κάτι που πάλι πάρα πολύ σωστή ρύθμιση. Ήδη βέβαια έτσι λειτουργούμε, άρα δεν θα αλλάξουν τόσο πολλά πράγματα. Δύσκολο να πούμε σήμερα τι σημαίνει αυτό όσον αφορά τις εξωτερικές υπηρεσίες. Όταν όμως διαβάζω αυτά τα λίγα έγγραφα που υπάρχουν, τότε καθησυχάζουμε. Ούτε η ΕΚΟ, ούτε οι συνεργάτες μας επιτόπου δεν πρόκειται να μπουν σε εξωτερικές υπηρεσίες. Αυτό με καθυσυχάζει. Γιατί έτσι μπορώ να καθισκάσω τους συνεργάτες μου, σταθερό του συστήματος, συνέχισε να δουλεύεις. Θα δουλεύεις όπου δουλεύεις και σήμερα. Άρα, εκεί, κάπως έτσι θα έχει το τελικό αποτέλεσμα. Τώρα, αν αλλάξουν τα πράγματα, τότε θα δούμε. Θα κάνω ό,τι μπορώ. Θα δω πώς μπορώ να αντιδράσω. Θα σας πω. Θα το κοιτάξω και θα σας πω. Μ' αρέσει ή δεν μ' αρέσει η εξέλιξη. Όμως, σήμερα όπως έχουν τα πράγματα δεν ανησυχώ. Impact Όμως, δεν θα υπάρχει τίποτα, μια τρομερή συνέπεια για τη δουλειά μας. Ας πούμε θα έχουμε τα γραφεία της ε, Επιτροπής και όπως είπαμε αν αλλάξει εκεί ο ιδιοκτήτης δεν θα αλλάξει η μίσθωση ας πούμε αν είναι πρόκειτο για, για μίσθωση. Τώρα Nous n'allons pas, Δεν μπορούμε να μπλοκάρουμε κάποια κεφάλαια, κάποιους πόρους, παρά το ότι θέλουμε να κάνουμε κάτι, αλλά όμως μόλις μπορέσει να υπάρξει κάποιο θετικό μήνυμα, σύμφωνα με το οποίο ε, θα φανεί κάποια στροφή στην κατάσταση, ξέρετε, η Γενική Διευθυνσή μας και με τη δική σας συνδρομή μπορούμε κάτι να κάνουμε. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι το δεν προβλέπονται κάποιοι κονδύλοι. δηλαδή σημαίνει δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Το ίδιο ισχύει και για το Πακιστάν. Το είχαμε 25 εκατομμύρια το 2010. Εάν κάτι χρειάζεται και μπορεί να γίνει θα το κάνουμε. Κάνουμε και παραπάνω. Τακτικά ενεργούμε κατά αυτόν τον τρόπο. Τώρα, όσον αφορά την αναθεώρηση του προγράμματος δράσης. Πρόκειται για σύστημα ευρείας συνένεσης. Πάμε για το πρώτο εξάμεινο του 2010. Και θα προχωρήσουμε με κάποια έκθεση πρωτοβουλίας και διαβούλευση επί της Βελγικής Προεδρίας. Και στην πορεία θα προσαρμοστούμε. Ε, ε, Τώρα όσον αφορά την υπερβολική βόσκηση αναφέρθηκε σχετικά με το τι γίνεται όσον αφορά τις περιοχές που από την ξηρασία όμως ίσως ο κίνδυνος είναι μικρότερος όπου έχουμε παραδοσιακές τεχνικές των τοπικών κοινοτήτων που είναι κάποιες οι οποίες δεν οδηγούν σε αυτό το φαινόμενο όπως στην Κένια. Εκεί έχει κάποιους ε, τείχους, κάποια, κάποια αναχώματα από την, ε, από την άμμο που φτιάχνουν ούτως ώστε να μην χύνεται το νερό και να αδειάζει ο μετροφόρος ορίζοντας. Όπως λέτε, επομένως αυτές οι παραδόσεις είναι βαθιά ριζωμένες εκεί και επομένως υπάρχει αυτή η απάντηση στο πρόβλημα. Τώρα, η μετάβαση, ούτως είπε, την ανθρωπιστική βοήθεια προς την ανάπτυξη στη Βόρεια Κένια. Εκεί ίσως θα καταφέρουμε, γιατί πρόκειται για μια περιοχή που, το λέω έτσι ανοιχτά μεταξύ μας, μην το πείτε στους Κενιάτες όμως, ότι δεν ενδιαφέρει